Κυρίε Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Κυρίσω την άναρξη της συνεδρίασής μας. Και πρώτα απ' όλα θέλω να καλωσορίσω θερμά εδώ τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όπως επίσης και τους συναδέρφους μας, ευρωβουλευτές. Θέλω ιδιαίτερα να χαιρετήσω τον κύριο Σορίν Λαζάρ, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Προϋπολογισμού και Τραπεζών, στην ε, Βουλή της Ρουμανίας, στο Κοινοβούλιο της Ρουμανίας, που θα κλείσει και τη σημερινή συνεδρίαση. Θέλετε μήπως και τώρα το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή ε, ευκαιρία που έχω να συμπροεδρεύω στο πλευρό σας σε αυτή τη συνεδρίαση. Θέλω να καλωσορίσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες και να τους ευχαριστήσω εξ ονόματος της χώρας μου, αλλά και προσωπικά για το ενδιαφέρον που δείχνετε για σημαντικά ευρωπαϊκά θέματα. Επίσης, ε, αυτό που μας ενδιαφέρει όλους είναι να βοηθήσουμε ε, την Ευρώπη να μεταξελιχθεί προς όφελος ε, των πολιτών μας. Καλωσορίζω αυτή τη συνεδρία στα πλαίσια της ε, Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας. Ήδη από την αρχή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το 2011 τα Εθνικά Κοινοβούλια είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν και να αυξήσουν το ρόλο τους για να υπάρχει μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση στη νέα οικονομική διακυβέρνηση και στη νέα αρχιτεκτονική. Ενισχύθηκε λοιπόν ο ρόλος των κοινοβουλίων και ελπίζω η παρούσα διάσκεψη να στεφθεί με επιτυχία. και περιμένω από τη συζήτηση να ακούσουμε νέες ιδέες και νέα επιχειρήματα, να ανταλλάξουμε απόψεις έτσι ώστε να ε, προωθήσει ε, αυτό την εκτέλεση του προπολογισμού και την κατάρτισή του γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτά τα ενθαρρυντικά λόγια, Πρόεδρε. Θέλω επίσης να καλωσορίσω εδώ και τα μέλη, του, τους βουλευτές από το Μαυροβούνι, την Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία, που είναι εδώ παρόντες και θα συμμετέχουν σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή η συνάντηση ε, με τους εθνικούς βουλευτές και τους ευρωβουλευτές για τον προπολογισμό. Γιατί αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, εσείς είσαστε αυτοί που ψηφίζετε τους πόρους από τον εθνικό Προϋπολογισμό κάθε φορά. Και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά ε, συζητάμε και ψηφίζουμε τις δαπάνες του ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Γιατί αντίθετα με τους εθνικούς βουλευτές, οι ευρωβουλευτές δεν έχουν ε, προνόμια. Οπότε εδώ το θέμα των ιδιών πόρων είναι η τελωνιακή δασμή... που όσο πάνε λιώνουν, εξατμίζονται όπως το χιόνι ε, στον ήλιο μετά από τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Η απόψενή συνεδρίαση θα επικεντρωθεί στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Γνωρίζετε ότι ε, ο ετήσιος προϋπολογισμός είναι δόση κάθε φορά ενός πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και τώρα η προγραμματική περίοδος αφορά το διάστημα 2014-2020. Είναι κομβική σημασία να συνεννοηθούμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Στις 14 Ενδεκάτου του 2018 το Κοινοβούλιο ενέκρινε την ενδιάμεση προσωρινή έκθεση για το τι μορφή θα πρέπει να έχει το πολιετε δημοσιονομικο δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 καθώς επίση και ήδη οι πόροι. Ήταν τη Επιτροπής Προπολογισμού. Η ενδιάμεση έκθεση αυτή βάζει ε, τι προτεραιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με συγκεκριμένα ποσά για ε, τι οροφές του PDP και για κάθε ε, τομεακό κλαδί δικό πρόγραμμα για την περίοδο πάντα 2021-2027. Τροποποιεί επίση τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρουσιάζει τι διεκδικήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα νέο σύστημα ιδίων πόρων. Ο προπολογισμό, το γνωρίζετε, αποτελεί και την έκφραση ενό οράματο. Εκφράζει μια πολιτική φιλοδοξία Και εμεί είμαστε υπεύθυνοι για να δώσουμε συνέχεια δεδομένων των δειγμάτων αναχρονισμού που βλέπουμε. Ο προπολογισμό λοιπόν πρέπει να είναι πιο απόλυτος αλλά και πιο κατανοητός για τους πολίτες. Οι νέοι μηχανισμοί εκτός προπολογισμού είναι κάτι που μπορεί κανείς να επικρίνει και νομικά μιλώντας, γιατί ουσιαστικά βραχυκυκλώνει την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ε, αρμόδιο σκέλος για τον προπολογισμό, αλλά και για τον έλεγχο. Έπειτα υπάρχει το θέμα της ενότητας επίσης του προπολογισμού και της διαφάνειας. Εγώ είχα φτιάξει ένα πίνακα που είναι ο γαλαξίας του προπολογισμού κατά κάποιο τρόπο και είναι ακριβώς το αντίθετο από τη διαφάνεια. Πρέπει λοιπόν να έχουμε στη διάθεσή μας τα μέσα να αντιδρούμε και στα πρόπτα. Στην εκτέλεση του δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2021 δεν είχαμε περιθώρια ελιγμών όταν προέκυψαν κρίσεις εκείνη ας πούμε της μαζικής μετανάστευσης του 2015. Ο προπολογισμό αυτός λοιπόν σήμερα αποτελεί το 1% του συνόλου των εθνικών ακαθάριστων εισόδων των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει την επιθυμία το κονδύλι αυτό να αυξηθεί κατά 30% και να είναι 1,3% το καθάριστο εθνικού εισοδήματος των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ή 28, ποιος ξέρει. Ποια θα είναι η σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση τους επόμενους μήνες ή χρόνια. 1,3% είναι αρκετά φιλόδοξο, είναι αλήθεια. Ε, πρέπει να πάμε όμως ακόμα πιο πέρα, αν θέλουμε η Ευρώπη να γίνει παγκόσμιο παράγοντας και αν θέλουμε να εξετάσουμε και να δούμε ποια είναι αυτά τα ευρωπαϊκά αγαθά που οι χώρες δεν ε, μπορούν να έχουν, δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν και να δούμε τι πιστώσεις μπορούν να πάνε υπέρ του ευρωπαϊκού προπολογισμού για να δείξουμε ότι έχουμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία αλλά πρέπει επίσης να συζητήσουμε τα επόμενα χρόνια ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στους δύο ειδικούς μας εισηγητές του πολιτούς δημοσιονομικού πλησίου. Ο κύριος Όλμπριχτ δεν μπόρεσε να έρθει, υπάρχει ένα πρόβλημα με το αεροπλάνο του και η κυρία το μας είναι άρρωστοι. θα αντικατασταθούν από τον κύριο Φερνάντες, που θα πάρει και το λόγο αυτής αμέσως, και στη συνέχεια η κυρία Καρδιά Ζαβάλα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαιρετίζω και εγώ εδώ όλους τους συναδέρφους, βουλευτές μπορούμε να μιλήσουμε για συναδέρφους, γιατί όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο, το καλό της Ευρώπης. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θέλω να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε δίκιο που ήθελε οι διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στην έκθεσή μου να είναι έτοιμο πριν από τις ευρωεκλογέ. Δεν τα καταφέραμε και δεν είναι δικό μας το σφάλμα. Εμείς είμαστε έτοιμοι, αλλά το Συμβούλιο για άλλη μια φορά δεν είναι έτοιμο. Και φοβάμαι ότι θα πάρει πολύ χρόνο και ο στόχος όλων των προγραμμάτων, όλων των συμφωνιών εταιρικής σχέσης θα ολοκληρωθούν ώστε να μπορούν να προχωρήσουν τα προγράμματα ε, τον Ιανουάριο του 2021. Αυτό θέλαμε, αυτό ήταν ο στόχο μας. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε και δεν φταίει το Κοινοβούλιο γι' αυτό. Επίσης, το Κοινοβούλιο ακολούθησε τη σωστή μεθοδολογία. Τη μεθοδολογία από κάτω προς τα πάνω. Τι κάναμε για να φτάσουμε στο 1,3% του καθάριστου εθνικού εισοδήματος. Κάναμε προσθέσει. Πολιτική συνοχής διατηρείται, κοινή γεωργική πολιτική, διατηρούνται οι άμεσες ενισχύσεις και η ανάπτυξη της υπαίθρου. Αλία, το ίδιο. Εράσμους συν, που αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις χώρες μέλη. Αυξάνουμε, τριπλασιάζουμε. Ο Ορίζον 2020, που τώρα ονομάζεται Ορίζον Ευρώπη, για την έρευνα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το πολυπλασιάζουμε επί 1,5. Χρειαζόμαστε επίσης ενίσχυση του Κοινωνικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για να βοηθήσουμε κυρίως τα παιδιά. 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει επίσης να διατηρήσουμε τις παραδοσιακές πολιτικές, όπως είπα, και ιδιαίτερα την πολιτική συνοχής. Ήταν απαράδεκτο να υπάρξουν περικοπές της τάξης του 40% στο Ταμείο Συνοχής. Επίσης, πολιτική άμυνας. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε έναν ευρωπαϊκό στρατό, αλλά θέλουμε να υπάρχει συντονισμός και θέλουμε εξοικονόμηση για να μπορέσουμε να έχουμε έρευνα και στην άμυνα. Και έχουμε και την ασφάλεια σε μια κατηγορία που είναι μεμονωμένη μόνη της για αυτό το στόχο. Φυσικά πρέπει να λυθούν και τα ζητήματα της μετανάστευσης. Οπότε προσθέτουμε την Ευρώπη 2020 στη στρατηγική της, την ενίσχυση των θεμάτων της μετανάστευσης και την ασφάλεια. Αλλά δεν είναι ένας ευρωπαϊκός στρατός όπως λένε μερικοί και νομίζουν ότι περί αυτού πρόκειται. Όχι. Οπότε Προσθέτουμε τα ποσά για όλες αυτές τις πολιτικές και το αποτέλεσμα είναι 1,3% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Με σταθερές τιμές. Και εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μερικές φορές μας μιλάει για σταθερές τιμές, κυρίως την πολιτική συνοχής, ενώ για την πολιτική γεωργική πολιτική στη χώρα μου μιλάει για τρέχουσες τιμές. Αλλά με τρέχουσες τιμές δεν βλέπουμε τις περικοπές, γιατί υπάρχει ο παράγοντας ε, πληθωρισμός. Για να μην υπάρχει σύγχυση λοιπόν, υπάρχει χωριστός πίνακας για μας τρέχουσες τιμές και χωριστός για σταθερές τιμές. Και θέλουμε να μιλάμε για σταθερές τιμές, γιατί εκεί φαίνεται ότι οι περικοπές είναι τεράστιες και απαράδεκτες στην πολιτική συνοχής. Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ικανή. Έχει τη δύναμη και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Και το Brexit δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη. Πρέπει να δείξει ακριβώς ότι είμαστε ικανοί και ότι θα πετύχουμε. Και γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε το 1,3%. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρέπει να το επενθυμίσουμε, είναι λιγότερο από το 1,1. Γιατί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, που ήταν εκτός προϋπολογισμού, τώρα συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοιες χειραγωγήσεις. Έχουμε μια εξαιρετική πρόταση. Τώρα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η πρόταση του Συμβουλίου. Ποια είναι αυτοί που θέλουν να κόψουν από την κοινή γεωργική πολιτική. Ποιες χώρες μέλη θέλουν περικοπές στην πολιτική συνοχής. Ποιος δεν θέλει να ενισχύσει την οικονομία ενισχύοντας το στόχο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και όλα τα οικονομικά και χρηματοδοτικά προγράμματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για αυτόν ακριβώς το στόχο. Πιστεύω λοιπόν ότι οι χώρες μέλη πρέπει να επιταχύνουν το ρυθμό. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αυτό που ξέρω είναι ότι τα άκρα της δεξιάς και της αριστεράς για άλλη μια φορά δείχνουν ότι είναι κατά. Καταψήφισαν και αυτή τη φορά, όπως πάντα. Είναι κατά του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, που είναι πολύ σημαντικό για τις επενδύσεις. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να ξεχνάει τις επενδύσεις, αλλά ούτε μπορεί να ξεχνάει την αλληλεγγύη. Και οι χώρες μέλη, το βλέπουμε, έχουν πρόβλημα μεταξύ τους. Είναι το πρόβλημα της εμπιστοσύνης που λείπει. Και εγώ θα ήθελα αυτή η εμπιστοσύνη μεταξύ τους να υπάρξει. Και επιμένω, όπως ξεκίνησε, εμείς είμαστε έτοιμοι, περιμένουμε και οι πολίτες και η Ευρώπη περιμένουν και αυτοί γιατί το χρειάζονται αυτό το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κυρία Καρτία Ζαμπάλ τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Ξανά βλέπουμε στο κοινοβούλιο μας τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προσπαθούν να συζητήσουν και να κάνουν διάλογο για το πώς πρέπει να είναι ο μελλοντικό προπολογισμό της Ένωσης. Τελειώνω από εκεί που τελείωσε ο Χωσέ, σταμάτησε ο Χωσέ Μαλουέλ είπε ότι ήμασταν έτοιμοι. Όντω, το Κοινοβούλιο είχε πει πω μία από τι προτεραιότητε τη θητεία αυτή ήταν η διαπραγμάτευση του δημοσιονομικού πλαισίου και σχεδόν όλη τη θητεία με αυτό το θέμα ασχοληθήκαμε. Τα πρώτα χρόνια είχαμε δώσει έμφαση στην αναθεώρηση του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, κάτι που μας επέτρεψε να δούμε ότι το πλαίσιο αυτό που είναι ένας επταετής προγραμματισμός είναι υπερβολικά άκαμπτο πλαίσιο δεν μας επιτρέπει να αντιδρούμε σε απρόπτες ε, εξελίξεις, σε κρίσεις που δεν έχουν προγραμματιστεί, σε ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί. Βασιζόμενοι σε αυτή την αναθεώρηση και μαθαίνοντας και από τα διδάγματα των ελλείψεων που διαπιστώσαμε για το υφιστάμενο πλαίσιο, ετοιμάσαμε μια νέα πρόταση για την περιοδο 2021 2021-2027. Όταν συναντηθήκαμε πέρσι, πάλι Φεβρουάριος ήταν, δεν είχαμε επιτάπητο στην πρόταση της Επιτροπής. Είχαμε όμως ένα σχέδιο του τι ήθελε να ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Κομισιόν. Μετά από πολλούς μήνες, χρόνια διαπραγματεύσεων, από αυτό που θέλαμε να ζητήσουμε στην Κομισιόν για το δημοσιονομικό πρέσιο και από αυτό που εν τέλει προτείναμε ως Κοινοβούλιο και ψηφίσαμε ως Κοινοβούλιο, με μεγάλη πλειοψηφία μάλιστα, δεν άλλαξαν πολλά. Ο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες εξήγησε ποια ήταν, ποιες ήταν οι προτάσεις μας. Υπογραμμίζω εκ νέου, διότι το θεωρώ σημαντικό, ότι οι προτάσεις αυτές εγκρίθηκαν με πολύ μεγάλη πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο, την πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων στο Σώμα, βουλευτές της αριστεράς, της δεξιάς, του βορρά, του νότου, της ανατολής, της δύσης, των πλουσιότερων και των φτωχότερων χωρών. Ήταν περίπλοκο. Το είδαμε στις διαπραγματεύσεις. Ήταν πολύ δύσκολο Χρειάστηκε σε κάθε περίπτωση μεγάλη συζήτηση μεταξύ μας για να φτάσουμε σε αυτή την κοινή πρόταση που όπως έλεγα προηγουμένως είναι 1,3% του ΑΕΠ της Ένωσης και είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε, το είπε και ο κ. Φερνάντες στην παρέμβασή του, ότι αυτό το νούμερο δεν είναι ένας ε, μαγικό αριθμός που έπεσε από τον ουρανό αλλά καπνό συζητήσεων, ανάλυσης επικοινωνίας και συζήτησης με τις εξειδικευμένες επιτροπές, διότι το δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είναι μόνο προπολογισμοί. Μιλούμε για προπολογισμού, αλλά προπολογισμού που πρέπει να χρηματοδοτήσουν ευρωπαϊκέ πολιτικές. Άρα με τους συναδέλφους από τις διάφορες εξειδικευμένες επιτροπές, περιφερειακή, γεωργίας, εξωτερικής, πολιτικής, ανάπτυξης, είδαμε ποιες πρέπει να είναι, ποιε είναι οι ανάγκης χρηματοδότησης της Ένωσης. Βέβαια, αφηρημένα, αν, το δει, αν δει κανείς ότι περνάει από το 1 στο 1,3% φαίνεται τεράστια η αύξηση, αλλά να θρήσουμε όλες τις ανάγκες που υπέδειξαν οι συνάδελφοι από τις επιτροπές και τις ε, προτεραιότητες που λέει το Συμβούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει στο μέλλον, το 1,3 ε, δεν έφτανε, θα έπρεπε να πάμε στο 2, στο 3%. Το 1,3 λοιπόν δεν είναι καρπός μεγάλων συζητήσεων μόνο, αλλά και καρπνό, καρπός περιστολής. Προχωρούμε με φιδό και παρότι θα μπορούσαμε κάλλιστα να ζητήσουμε 2 ή 3% του ΑΕΠ, έχουμε επίγνωση ότι αυτή τη στιγμή μια τέτοια συζήτηση δεν μπορεί να γίνει. Το 1,3 λοιπόν είναι το άθροισμα των ελάχιστων αναγκών που η Ένωση πρέπει να καλύψει τα επόμενα έτη. Και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό συχνά. Όταν μιλάμε για προπολογισμό ακούγεται η φράση να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Δεν γίνεται αυτό. Αν θέλουμε να υλοποιήσουμε τι προτεραιότητε μα δεν μπορούμε να το κάνουμε με λιγότερα χρήματα. Θέλουμε μεγαλύτερη, περισσότερη άμυνα, πρέπει να δώσουμε περισσότερα κονδύλια. Αν θέλουμε μια πολιτική υποδοχή προσφύγων και διαχείριση των εξωτερικών κοινών μα συνόρων, χρειαζόμαστε περισσότερου πόλους. Αν θέλουμε να κρατήσουμε τη γεωργία στα επίπεδα που έχουμε τώρα ή να αναπτύξουμε τι περιφερειές μα, δεν μπορούμε να περικόψουμε τα ευρωπαϊκά αυτά προγράμματα. Και πρέπει να είμαστε σαφείς. Το Κοινοβούλιο έχει μία πλήρη, ξεκάθαρη θέση και θέλουμε να ξέρουμε και τη θέση του Συμβουλίου στο σημείο αυτό, γιατί συχνά το Συμβούλιο λειτουργεί ως Ιανός και το συζητούμε αυτό στο Κοινοβούλιο. Κάθε φορά που έχει Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εμφανίζονται νέες προτεραιότητες, νέες ανάγκες, εμφανίζονται νέες πολιτικές. Την ώρα της αλήθειας όμως δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε. Χωρίς νέα κονδύλια, τι νέες πολιτικές μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Αν θέλουμε νέες πολιτικές, θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια αύξηση. Δεν θα μπω στα θέματα των ίδιων πόρων που είναι άλλοι συνάδελφοι που θα το σχολιάσουν. Ένα τελευταίο σχόλιο. Οι διαπραγματεύσεις για το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι περίπλοκες διότι υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις δουλειάς. Η μία είναι η καθαρά δημοσιονομική, το πλαίσιο. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και τα το νομοθετικό κανονισμό και την έκθεση για τους ίδιους πόρους. Αυτά τα τρία σκέλη δεν μπορούν να δουλευτούν ξέχωρα. Δεν μπορούμε να ορίσουμε πολιτικέ χωρί χρήματα, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσα χρήματα θα χρειαστεί μια πολιτική αν δεν έχουμε σαφή την πολιτική και προφανώ χρειαζόμαστε να ξέρουμε πώ θα τι χρηματοδοτήσουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν θεωρεί θεμελιώδες να μπορεί να δουλέψει παράλληλα και στους τρεις, στα τρία αυτά σκέλη της δουλειάς. Δημοσιονομικό πρέσιο, τομεακοί προπολογισμοί και ήδη πόροι. Και θα το κάνουμε με όλη τη δυνατότητα συνεργασίας που ελπίζουμε να λάβουμε από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από το Συμβούλιο και την Προεδρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ίντερ. Ευχαριστώ. Ακόμα πιο δύσκολο να συζητήσουμε με το Συμβούλιο. Καθή στιγμή η εντολή που έχει να δώσει το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα. Σας αφήνω να φανταστείτε τις σκληρές συζητήσεις στο Συμβούλιο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γιάννος Λεβαντόφσκι για τους ιδίους πόρους. Όχι. Ε, πώς θέλετε. Ε, good afternoon. Welcome to, to... Ε, γεια σας. καλώ ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα αρχίσω από ένα γενικότερο σχόλιο. Πώς σχεδιάζει κανείς και πώς διαπραγματεύεται το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι από τις πιο καθοριστικές στιγμές της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αφορά το μέλλον σε αριθμούς αυτούς. Δεν είναι απλή διακήρυξη αλλά ο προϋπολογισμός είναι το ίδιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι κούφια λόγια. Και αυτό αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει τίποτα αντίστοιχο ε, στους εθνικούς προϋπολογισμούς που έχουν ενιάψιο χαρακτήρα. Εμείς έχουμε πολιετής προϋπολογισμούς, επενδυτικούς και οι επενδύσεις ε, κατά κανόνα και κατεξοχή είναι πολιετής. πάντα υπάρχουν ειδικέ περιστάσεις, γι' αυτό τσακώνονται τα κράτη-μέλη. Ποτέ δεν είναι τα πράγματα κανονικά. Τα έχω ζήσει και παλαιότερα. Το 2005, το 2006 ήταν το Big Bang της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διεύρυνση δηλαδή, αλλά μπήκανε 10 καθαροί αποδέκτες και καθένας καθαρός συνεισφορέας το 2004. Το 2011 με 2013 το θέμα ήταν ε, η βαθιά κρίση και το πρόβλημα ε, του Brexit τότε και ο κύριος Κάμερον που προετοίμαζε το δημοψήφισμα και τώρα έχουμε το Brexit και ε, ε, πιέσεις να υπάρχει ένας ειδικός προπολογισμό για τις χώρες της Ευρωζώνης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βοήθησε πάρα πολύ να ολοκληρωθεί η συμφωνία πριν τις ευρωεκλογέ, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία άνοιξαν ε, τους λεγόμενους εθνικούς φακέλους οι εμπειρογνώμονες ε, εύκολα υπολογίζουν τι σημαίνει αυτό για την Πολωνία, για την Πορτογαλία ε, ε, και το, το κάνουν. Αλλά για πρώτη φορά αυτό δημοσιεύθηκε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι κάποιες χώρες θα χάσουν 24-25% της χρηματοδότησης και άλλες θα κερδίσουν. Δεν βοηθάει πάρα πολύ αυτό στην επίτευξη συμφωνίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ακούσαμε, έχει πάρει θέση για πρώτη φορά και με ποσά, αλλά δεν τρέφει καμία αυταπάτη ότι θα ολοκληρωθεί η προσπάθεια αυτή, δεν θα προλάβουμε πριν τις ευρωεκλογέ. Ε, την περασμένη φορά ήμουν αρμόδιος επίτροπος και χρειάστηκαν δυόμιση χρόνια για να συμφωνηθεί. Τώρα φανταστείτε ε, να προλάβουμε πριν τις ευρωεκλογέ να συμφωνήσουμε. Σε ό,τι αφορά <clears throat> τα έσοδα, είμαστε εισηγητές για το κοινοβούλιο μαζί με το Gérard Ντεπρέ που μπορεί να είμαστε από διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις, αλλά μιλούμε με μία φωνή. Που είναι παράδοξο, γιατί υφίσταται πολλές ε, κριτικές ε, ο κλάδος των εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αλλά γενικά είναι στάσιμος και σταθερός από το 1988 και πραγματικά θα πρέπει αυτό να πιστωθεί στους Βρετανούς γιατί οι Βρετανοί περασπίστηκαν την Βρετανική επιστροφή, το rebate, έγιναν κάποιες διορθώσεις και κάποιες προσαρμογές και μετά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει το σύστημα. Παρόλο που δεχόταν όλη αυτή τη σκληρή κριτική ότι είναι κατανόητο για τον κόσμο και αδιαφανές το σύστημα των εσόδων. Τελευταία απόπειρα ήταν η δική μου ε, για να επιβάλλω το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και βελτιωμένο ΦΠΑ, αλλά το απέκρουσε γρήγορα ο κύριος Κάμερον. Και τώρα το Brexit δεν είναι πρόβλημα, είναι μια ευκαιρία να εξυγχρονιστεί ε, το σκέλος των εσόδων του προπολογισμού. Γι' αυτό έχουμε κάνει τη μετεοπαθή αυτή και προσεκτική πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 12% του συνόλου των εσόδων θα προέρχεται από τους νέους ιδίους Η κοινή ενοποιημένη βάση για τη φορολόγηση ε, των ε, εταιριών, ε, τα πλαστικά, τα μη ανακυκλούμενα και ο μόνο φόρο που είναι δημοφιλή είναι ο φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Γιατί τιμωρεί τι τράπεζε που ευθύνονται για την οικονομική κρίση. Ε, αυτό που δεν μου αρέσει ε, στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι από την αρχή έγιναν κάποιε διορθώσει ε, για την Αυστρία, για τη Δανία, για τη Γερμανία και για τις κατοχώρες. Συνήθως αυτές οι διορθώσεις ε, είναι ένα δώρο που γίνεται τελευταία στιγμή, την τελευταία νύχτα κιόλα ε, στις χώρες που είναι καθαροί οι συνεισφορείς. Τώρα το είχαμε από την αρχή. Η θέση του Κοινοβουλίου ποια είναι. Και θα πρέπει να το λέμε ξεκάθαρα ότι εμείς είμαστε εκλεγμένοι βουλευτές από τις 28 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε απολύτως υπέρ της φορολογικής, της δημοσιονομικής κυριαρχίας των κρατών μελών. Οι αποφάσει για του ιδίους πόρους θα πρέπει να λαμβάνονται ομόφωνα και να κυρώνονται από τα εθνικά κοινοβούλια. Και σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούμε τη φορολογική και την δημοσιονομική κυριαρχία των κρατών μελών. Ε, ποιο είναι το καινούριο, ένας νέος ίδιος πόρος. Ε, είναι κάτι που θα μειώσει την εισφορά του ΑΕΠ των κρατών μελών, που το 80% και πάνω ε, είναι από το ΑΕΠ των κρατών και είναι καλό σταθεροποιητή γιατί είναι το πιο προβλέψιμο σκέλος εσόδων. Γιατί όμως να μην προσπαθήσουμε να βρούμε ε, ένα κλάσμα ε, όχι νέων φόρων, αλλά κείμενο, υφισταμένων φόρων, ας πούμε της φορολόγησης των επιχειρήσεων. Μπορούμε να βγάζουμε κάποια χρήματα για το ευρωπαϊκό σύστημα εκπομπών, δεν είναι και καμιά επανάσταση. Εγώ έχω περιορισμένες προσδοκίες δεδομένης της εμπειρίας μου. Υπάρχουν κάποιες χώρες που τα έχουν στυλώσει από την αρχή σε οποιοδήποτε εξυγχρονισμό του συστήματος των ιδίων πόρων. Ο άλλος είναι πιο πρόθυμες. Υπάρχει κάτι που λέγεται ε, απλουστευμένες διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο. Δεν είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά αυτά που ακούμε. Υπάρχει όμως μια ευκαιρία. Ε, ε, Μέχρι τώρα λοιπόν η Μεγάλη Βρετανία ήταν εκείνη που κρατούσε έτσι, σε αυτά τα σταθερά επίπεδα τα έσοδα. Τώρα υπάρχει κάποια ελπίδα να εξυγχρονιστεί το σύστημα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννος. Ο κύριος ο άλλος εισηγητής για τους ίδιους πόρους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, θέλω να πω δύο λόγια μετά τον συνάδελφο Λεβαντόφσκι. Στις ε, συζητήσεις που ξεκινούμε να έχουμε τώρα, εν ώψη των επόμενων ευρωεκλογών, υπάρχει κάτι που μας λέει ο κόσμος. Φοβούνται Ευρωπαϊκό Φόρο. Το πρώτο που θέλω να πω εγώ είναι ότι στους ίδιους πόρους που εμείς προτείνουμε δεν υπάρχει ευρωπαϊκός πόρος. Δεν είναι πρόταση επιτροπής που θα εγκρίνει το Κοινοβούλιο. Η φορολογική κυριαρχία, η δημοσιονομική κυριαρχία των χωρών μελών παραμένει. Για να υπάρξει συμφωνία για τους ίδιους πόρους πρέπει να υπάρξει απόφαση από το Συμβούλιο με ομοφωνία βάσει πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από απλή γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν έχουμε δηλαδή καμία απολύτως εξουσία πάνω σε αυτό. Είναι στα χέρια των χωρών μελών που μπορούν να πούνε ναι ή όχι στην επικύρωση του κάθε ίδιου πόρου. Και γιατί το λέω αυτό γιατί εδώ υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις με την κοινή γνώμη και μας κατηγορούν για τα χειρότερα κακά. Δεύτερον, το σύστημα ιδίων πόρων που προτείνουμε εμείς και που το παρουσίασε κάπως ο κ. Λεβαντόφσκι, δεν έχει σαν στόχο να αυξήσει την δημοσιονομική και φορολογική πίεση. Οι ίδιοι πόροι προοδευτικά θα τροφοδοτούν όλο και περισσότερο τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για να μειωθεί η συνεισφορά των χωρών μελών. Και γιατί το θέλουμε αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι ότι από τον εθνικό προπολογισμό ο καθένας ε, τα μετράει και λέει ορίστε εγώ τόσα έβαλα στο ταμείο, τι πήρα πίσω. Είναι αυτή η νοτροπία της δίκαιας επιστροφής που έχει γενικευθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν οι εκείνοι οι οποίοι είναι καθαροί εισφορείς και εκείνοι οι οποίοι είναι καθαρά αποδέκτες. Το κοινό συμφέρον των Ευρωπαίων, δηλαδή, τελικά, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Και σε πρώτη μοίρα μπαίνει το τι βάζω, τι παίρνω. Κάτι άλλο που αιτιολογεί την εισαγωγή των ε, ιδίων πόρων είναι ότι θα υπάρξει μία τρύπα με την έξοδο των Βρετανών που είναι 13-14 περίπου εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό. Ορισμένες χώρες βρίσκονται σε κάπως ε, λεπτή θέση δεδομένου του χρέους τους και θα περάσει κάτι τέτοιο στη κοινή γνώμη ότι πρέπει να πληρώσουν οι άλλοι για την αποχώρηση των Βρετανών. Τώρα αν θέλουμε να πετύχουμε την ισορροπία που προβλέπεται στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως τα παρουσίασαν ο Χωσέ Φερνάντες και η Γκαρδία Σαμπάλ, αν θέλουμε τέτοια δημοσιονομική ισορροπία, δεν είναι δυνατόν να βρούμε χώρο για τις νέες προτεραιότητες και όλα να τα φορτωθούν οι εθνικοί προπολογισμοί. Εξού και εμείς προτείνουμε πρώτα απ' όλα όχι μόνο έναν πόρο, ένα πακέτο νέων ε, πόρων. Γιατί ώστε η συνεισφορά να μην είναι δυσανάλογη. Αν, ας πούμε, υπάρχει ο ΦΠΑ, υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες θα συνεισφέρουν περισσότερο από άλλες. Αν σε αυτό βάλουμε και ένα δεύτερο ιδιοπόρο, ας πούμε, μια εισφορά στο σύστημα εκπομπών, μπορεί να εξισορροπήσετε εν μέρη, αν προσθέσετε και ένα τρίτο στοιχείο. Την φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα υπάρξει πάλι εξισορρόπηση. Προτείνουμε λοιπόν ένα πακέτο έτσι ώστε ακριβώς να μπορεί να υπάρξει εξισορρόπηση στις συνεισφορές των χωρών μελών και να είναι δίκαιο το σύστημα βάσει του εθνικού πλούτου. Και το τελευταίο, εμείς δεν λέμε ότι όλοι οι ίδιοι πόροι πρέπει να εισαχθούν συγχρόνως από 1η Ιανουαρίου 2021 ένα πακέτο δύο πόρων το οποίο θα είναι ξέρω 15 δισεκατομμύρια, 20-30 νέοι ήδη πόροι. Όχι. Αν όπως το πρότεινε ο κύριος Λεβαντόφσκι έχουμε μια κάποια εισφορά για τον, τη φορολογία εταιριών, ήδη κάτι θα είναι. Πρέπει να συμφωνήσουμε δηλαδή πρώτα για την κοινή ενωπημένη βάση φορολογία εταιριών και μετά να δούμε πώς αυτή θα συμπεριληφθεί στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ο μηχανισμός λοιπόν που προτείνουμε εμείς, αν μπορώ να το συνοψίσω με δύο λόγια, είναι να επιτρέψουμε μια μείωση των συνεισφορών με τη βοήθεια ενός πακέτου ισορροπημένου νέων πόρων που θα επιτρέπει να χρηματοδοτήσουμε και την αποχώρηση των Βρετανών και νέες προτεραιότητες που διατυπώνονται στον προπολογισμό και έχουν ήδη εντοπιστεί. Έρευνα, καλύτερος έλεγχος των συνόρων μας, μεταναστευτικό, ζητήματα σημαντικά και σημασία τους, παρά το ότι πιστεύουν ίσως κάποιοι, θα αυξηθεί στο μέλλον και δεν θα μειωθεί. Τίποτα δεν θα σας επιβληθεί αν δεν το ψηφίσετε. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα ήταν καλό να έχουμε νέους ίδιους πόρους και έχουμε εμπιστοσύνη στα Εθνικά Κοινοβούλια να καταλάβουν την επιχειρηματολογία μας. Αν δεν συμφωνήσουμε μαζί για το κοινό ε, καλό, αν παραμείνουμε στο πόσα βάζω, πόσα παίρνω, υποθηκεύουμε την ίδια την έννοια της αλληλεγγύης και δεν θα λύσουμε κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ζεράρ. Βλέπετε συνάδελφοι πόσο στην πράξη πρέπει να τετραγωνίσουμε τον κύκλο για να λύσουμε το πρόβλημα. Πρέπει με περιορισμένα μέσα να λειτουργήσουμε αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις, μετανάστευση, άμυνα, κλίμα, ψηφιακή οικονομία. Είναι εντυπωσιακό το ότι ούτε ένας γίγαντας της ψηφιακής οικονομίας δεν είναι στην Ευρώπη. Έχουμε ίδιους πόρους που είναι εξαιρετικά περιορισμένοι, 10%, του προπολογισμού. Το 90% προέρχεται από τα κράτη-μέλη. Είναι εισφορές που εντάσσετε εσείς ε, στους εθνικούς σας προϋπολογισμούς. Όταν λέμε λοιπόν ότι μπορούμε να ανεβάσουμε τον προϋπολογισμό στο 2-3% αυτό θα πρέπει να γίνει χωρίς ε, αύξηση των δημοσίων δαπανών στην Ευρώπη. Να μπορείτε δηλαδή να αναδείξετε να, μειώ, να αξιολογήσετε κάποιες εθνικές δαπάνες και να δείτε αν ε, ανταποκρίθηκαν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και αν φαίνεται ότι σε κάποιους τομείς θα μπορούσαμε να δαπανούμε πιο χρήσιμα τους πόρους που, έχουν, που δεσμεύονται σε εθνικό επίπεδο, σε μια τέτοια φάση είναι δυνατό να μεταφέρουμε στον ευρωπαϊκό Προπολογισμό εθνικές δαπάνες όσο αυξάνεται ο εθνικό προπολογισμό πρέπει να μειώνεται τα ποσά των εθνικών προπολογισμών Τούτου λεχθέντος. Θα σα δώσω το λόγο αγαπητοί συνάδελφοι. Να πω καταρχάς ότι θα δώσουμε το λόγο στους, σε όσο περισσότερου από εσά θέλετε να μιλήσετε. Σα καλώ να συμπληρώσετε αυτές τις κάρτες που έχετε μπροστά σας να τα δώσετε στους κλητήρες ε, στην αίθουσα που θα το μεταφέρουν σε εμά. Θα, το θα δίνω το λόγο σε δύο εθνικούς βουλευτές, ο τρίτος θα είναι ευρωβουλευτής και ούτω καθεξής. Θα δούμε αν χρειάζεται να μειώσουμε το χρόνο ομιλία. αλλά αν μπορείτε να μιλήσετε δύο λεπτά, τρία το πολύ, θα μιλήσουν όλο όσο περισσότερο γίνεται. Δίνω αμέσως το λόγο. Στην κυρία Νέτ Μπόσα. Madame Bossa. Good afternoon to everyone. I would like to... Καλησπέρα. Θα μιλήσω ουγγρικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πάρω το λόγο. Ήθελα να πω ότι είναι ιδιαίτερα θετικό και η Ένωση να υποστηρίζει την καινοτομία και να μπορούμε έτσι να αντιμετωπίσουμε καλύτερο, καλύτερα τον 21ο αιώνα. Αυτό είναι καθοριστικό για τι πρέπει να ζήσουμε σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι Παρά την παγκοσμιοποίηση υπάρχουν χώρες και περιφέρειες που χρειάζονται ιδιαίτερους πόρους για να αναπτυχθούν ακόμα και σήμερα. Με τους πόρους αυτούς θα δημιουργήσουμε μία κοινότητα, μία, ένα ισχυρό ε, συνδετικό κρίκο. Αυτό είναι το απαιτούμενο. Δεν το λέω αυτό γιατί θέλουμε να είμαστε καθαροί δικαιούχοι, γιατί θέλουμε περισσότερα χρήματα, αλλά γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει εδώ για να βοηθήσει αυτόν που έχει ανάγκη να αναπτυχθεί. Μόνο έτσι πιστεύω μπορούμε να μείνουμε να παραμείνουμε μια κοινότητα ελευθερίας και ελεγγύης και μόνο έτσι δεν θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαφυλάξει αλλά και να ενισχύσει την θέση της στην παγκόσμια οικονομία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να, να... επανέλθουμε σε αυτές τις σκέψεις. Η πόρη για τη συνοχή θα αποτελούσαν μια θετική συμβολή αν καταλάβαιναν και αυτούς που ζητάνε τις ανάγκες αυτές. Ο κύριος Ντόρατε Πατσέκο από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. <laughs> Ευχαριστώ. Καταρχήν, εξ ονόματος του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου θέλω να δηλώσω ότι είμαστε υπέρ της ενίσχυσης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε όμως, συχνά λέμε ότι μελέτα κάνεις μόνο σπάζοντας αυγά. Δεν μπορεί να κάνεις ομελέτα χωρίς αυγά. Αν θέλεις λοιπόν νέους κλάδους παρέμβασης της Ένωσης πρέπει να τους χρηματοδοτήσεις. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε λοιπόν την παράμετρο έσοδα. Είναι σημαντικές οι πολιτικές, ε, απαιτούν, ε, είναι σημαντικές οι ικανότητες καινοτομίας που έδειξε η Επιτροπή που δεν περιορίστηκε στις παραδοσιακές πολιτικές για να είναι πιο ανταγωνιστικός ο ευρωπαϊκός χώρος στον κόσμο. Τούτος δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν υπονομεύοντας τις πολιτικές συνοχής, ωστόσο. Ε, είπε και η Ρουμανική Προεδρία ότι οι πολιτικές συνοχής είναι καθοριστικές. Μίλησε υπέρ της Ευρώπης της σύγκλησης. Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η μείωση των ανισοτήτων ανάπτυξης και να προσφέρουμε όλες τις δυνατότητες ε, σε όλους τους πολίτες της Ένωσης για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Είμαστε λοιπόν όλοι υπέρ της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να αναπτυχθεί αυτός ο χώρος διαλόγου. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να γνωρίζει ότι έχει την υποστήριξη των Εθνικών Κοινοβουλίων στην μεγιστοποίηση του προπολογισμού της Ένωσης για νέες πολιτικές, αλλά και για την ενίσχυση της πολιτικής σύγκλησης σε έναν ευρωπαϊκό χώρο που είναι το θεμέλιο αυτό που ήθελαν οι ιδρυτικοί πατέρες τη Ένωσης. Αυστρία. Ο κύριο Ρούμπιγκ, Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Το μέλλον τη Ευρώπη εξαρτάται από τρία μεγάλα θέματα ουσιαστικά. Και πιστεύω ότι ένα από τα σημαντικότερα είναι η προστιθέμενη αξία που φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί Πραγματικά κάνει τη διαφορά αυτό. Άλλο είναι να κάνει ε, κάτι μία χώρα μόνη της και άλλο να τα κάνει μαζί με 27 άλλα κράτη. Και αυτό επιβαρύνει και το φορολογούμενο. Εκεί αν προωθούμε εκείνα τα προγράμματα και τις πολιτικές όπου υπάρχει πραγματικά ευρωπαϊκή υπεραξία ή προστιθέμενη αξία. Και το δεύτερο είναι τι κοστίζει στους πολίτες. Ε, έλλειψη ευρωπαϊκής συνεργασίας, το κόστος της μη Ευρώπης, αν θυμάστε, θα πρέπει να το υπολογίσουμε, όπως και την προστιθέμενη αξία. Γιατί αυτοί οι δύο πυλώνες ουσιαστικά μας εγγυώνται ότι ε, θα φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πολίτες. Και τρίτο στοιχείο είναι η αρχή της επικουρικότητας. Θα πρέπει ο κάθε πολίτης να αποφασίζει ό,τι μπορεί ο ίδιος και όσα μπορεί και μετά το αμέσως επόμενο επίπεδο να τον βοηθάει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είμαι εγώ εδώ παλιά καραβάνα, στην τελευταία δέκα πενταετία έχουμε δει ε, από το ένα 0,12% ε, του ΑΕΠ να γίνεται η συνεισφορά 0,9% ε, στον προπολογισμό του 2019. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι <coughs> μαζί με τον Πρόεδρο Αρτοή ότι καταφέραμε το τρομακτικό κατόρθωμα 0,9%. Από το 1,12 έχουμε πάει ε, στο 0,9. Και ετησίως 1% ε, των θέσεων των υπαλλήλων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν περικοπεί και 4% του συνόλου των ε, διοικητικών δαπανών. Άρα, αφού συζητάμε τώρα για τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν οι παραδοσιακές δαπάνες που χρειάζονται κάποια αναπροσαρμογή, να θέσουμε νέα κέντρα βάρους, περισσότερο στην έρευνα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτές πληρώνουν τους περισσότερους φόρους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μια κοινωνική Ευρώπη. Ότι εκείνοι που πληρώνουν τους περισσότερους φόρους να υποστηρίζονται για να μπορούν να τους καταβάλουν. Και για την νεολαία μας το πρόγραμμα Erasmus Συν. Αυτά είναι τα σημαντικά. Στα σημαντικά θα πρέπει να επικεντρωθούμε και μετά να δούμε και ποιες είναι οι νέες ευθύνες που καλείται και οφείλει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, προ όφελο των πολιτών. Και το ε, ένα αυτό εκατό που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας, κανονικά θα πρέπει να συμφωνηθεί ε, ότι είναι η οροφή για τις παλιές υποχρεώσεις. Αν έχουμε νέες υποχρεώσεις, χρειάζονται και περισσότερα χρήματα. Έχοντας υπόψη τα τρία προηγούμενα που είπα, το κόστος της μη Ευρώπης, την επικουρικότητα και την προστιθέμενη αξία για να εργαζόμαστε πάντα προς το συμφέρον των πολιτών. Ευχαριστώ, Πάουλ. Ευχαριστώ. Από την Γερμανική Βουλή, Bundestag από την Επιτροπή Προπολογισμών, μουρμουρίζει ο Πρόεδρος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω δύο λόγια για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα είχα να πω πάρα πολλά, αλλά επειδή δεν έχω χρόνο θα περιοριστώ. Το μεσοπρόθεσμο, ε, τι είναι, η πολιτική που έχει ε, σφυριλατηθεί σε ποσά. Εσείς το είπατε τετραγωνισμό του κύκλου, εγώ θα το έλεγα συμβιβασμό. Ορισμένοι προλαλήσαντες εξήγησαν τις διαδικασίες που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να αυξηθούν οι συνεισφορές. Ε, είπατε ότι γίνανε προτάσεις από τη βάση προς την κορυφή. Ε, Εμεί στη Γερμανία έχουμε ε, τα τελευταία χρόνια κάνει ε, μια καλή εμπειρία ε, με την αντίστροφη διαδικασία top-down, όχι bottom-up. Και ε, πρέπει να κλείσουμε δύο ελλείμματα το Brexit γιατί φεύγει ένας καθαρός συνεισφορέας και οι δεύτερες νέες προκλήσεις όποιες και αν είναι αυτές έρευνα, ψηφιοποίηση, νεολαία προστασία του κλίματος ακούστηκαν μετανάστευση, προστασία των συνόρων ασφάλεια και άμυνα με τις διάφορες πτυχές τους αλλά το θέμα είναι πάντα που βρίσκεται η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για να ε, παραχθεί χρήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Συμβιβασμός θα είναι για να κλείσουν αυτές οι δύο τρύπες, ε, ε, συνδυασμός περικοπών και νέων δαπανών αλλά είναι τα συμφέροντα που θα συγκρουστούν διαφορετικά. Ε, μπορεί να είναι Ανατολή-Δύση ή Ανατολή-Νότος, Βορράς-Νότος, ε, συνεισφορή, καθαρή Όλοι θα πρέπει να κάνουμε υποχωρήσεις. Στη Γερμανία θα κάνουμε περικοπές. Ε, ανησυχούμε πολύ για τη Γεωργία, αλλά ακόμα και αν κάνουμε περικοπές στη Γεωργία και πάλι σε κάποιους τομείς θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε αν υπάρχει ασφάλεια προγραμματισμού για μια επταετία που είναι και η προγραμματική περίοδος για να μπορεί ο καθένας να κανονίζει την πορεία του για το επόμενο διάστημα. Ισορροπία μεταξύ των παλαιών και νέων ευθυνών, προτεραιότητες πρέπει να ορίσουμε και κυρίως ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης, πόσο αξίζει για μας η Ευρώπη να βάλουμε ένα σύνολο προϋποθέσεων και κανόνων που ενδεχομένως να προσανατολίσουμε σε αυτούς και ε, τη χρηματοδότηση. Και αν θέλουμε να διαπραγματευόμαστε επί ώρε ώρες με την Κίνα, με τι Ηνωμένε Πολιτείε, θα θέλουμε αποτελέσματα, αν θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή των Ευρωπαίων σε ένα καλύτερο περιβάλλον, ε, μόνο από κοινού θα τα καταφέρουμε. Καμία χώρα δεν μπορεί να το κάνει από μόνη τη. Καμία χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζω μέχρι το φθινόπωρο να έχουμε καταλήξει για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Μαργαρίτα Μάρκουες. Πορτογαλία. Εκτός μικροφώνου, δεν ακούγεται. Δεν δουλεύει το μικρόφωνο της ομιλήτριας μάλλον. Δυστυχώς δεν ακούγεται. ça marche. Τώρα είναι εντάξει. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Προπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει βάλει το θέμα αυτό στην εμερήσια διάταξη της κοινοβουλευτικής αυτής της εβδομάδας. Είναι πολύ σημαντικό για μας τα Εθνικά Κοινοβούλια που και εμείς συζητάμε για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο δημιούργησε μία ειδική επιτροπή για να μας συνοδεύσει σε αυτήν την προσπάθεια της συζήτησης για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και ο κύριος Αρτουή, ο πρόεδρος Αρτουή είναι ακριβώς ένας, μία από τις προσωπικότητες που προσκαλέσαμε σε ακρόαση στην επιτροπή αυτή. Και μεθαύριο θα συζητηθεί το θέμα στην Ολομέλεια του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου. Εγώ εισηγήτρια εκ μέρου των σοσιαλιστών. Θέλω επίσης εδώ να αναγνωρίσω και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη προηγούμενη εβδομάδα, που αποφάσισε να αντιταθεί στην μείωση των κονδυλίων για την πολιτική συνοχή και για την μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Είναι δύο στοιχεία πολύ σημαντικά αν θέλουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να λειτουργήσει ικανοποιητικά. Έχω τώρα μερικές παρατηρήσεις σύντομα. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν αρκετά φιλόδοξη όσον αφορά τους ίδιους πόρους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ευκαιρία να επιδείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία. Δεν το έκανε όμως. Και ακόμα και για την συμμετοχή του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Ο Υπουργός στην Πορτογαλία είχε πει ότι μπορούσε να συζητήσει μεγαλύτερη συνεισφορά από πλευρά τη Πορτογαλίας, υπό κάποιους όρους βέβαια, προκειμένου να φτάσουμε στο 1,3% που είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θέλω να έρθω και σε δύο προτάσεις για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα έπρεπε να προστατευτούν. Πρώτον, δημιουργία ενός μηχανισμού στήριξης των μεταρρυθμίσεων στις χώρες μέλη. Και δεύτερον, ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα για τι επενδύσει. Αυτά τα δύο στοιχεία πρέπει να τα φροντίσουμε πολύ και να τα προστατεύσουμε στι διαπραγματεύσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δυσκολευτεί να εγκρίνει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάτι το οποίο ε, κινδυνεύει να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, αν περιμένουμε το επόμενο κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό η αρχή ε, νη συνπρία να διατηρηθεί και να εξετάσουμε όσο γίνεται περισσότερο χωρίς προβλήματα να προχωρήσουμε και χωρίς διακοπές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Ουλέινεν από την Πούντεστακ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω ότι φυσικά ο προπολογισμό και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή ιδέα, το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Και φυσικά δεν έχει να κάνει μόνο με τους ιδίους πόρους και τα οικονομικά. Ε, ε, θα πρέπει να μας απασχολήσουν αυτά και να μας προβληματίσουν, αλλά το κυριότερο δεν είναι για μας το ποσό ή το ποσοστό 1,1 ή 1,3 όπως επιθυμείτε εσείς για τους ίδιους πόλους. Για μας αυτό που είναι προφανές και αυτονόητο είναι να καθίσουμε, να κοιτάξουμε και να αξιολογήσουμε το σκέλος των δαπανών και να κοιτάξουμε εάν όλα αυτά που κάνουμε μέχρι τώρα είναι απαραίτητα και στο μέλλον. Ε, τηρείται πάντα η αρχή της επικορικότητας είναι σκόπιμα όλα αυτά τα έξοδα. Δηλαδή να μην κοιτάμε μόνο τα έσοδα αλλά και τα έξοδα. Ε, να βάλουμε λίγη τάξη αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Ε, βέβαια, το είπαν ήδη πολλοί συνάδελφοι, θα πρέπει να κοιτάξουμε ότι σε κάποιους ε, τομείς μπορεί να χρειαστούν περικοπές και συμβιβασμοί με ε, παραχωρήσεις και στη γεωργική πολιτική. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον συνάδελφο. Στη Γερμανία βέβαια αυτό θα μας πονέσει πολύ. Αλλά στο δεύτερο πυλώνα της κοινή γεωργικής πολιτικής θα μπορούσε να γίνει αυτό. Αλλά έχουμε προτεραιότητες όπως είναι η παιδεία, η έρευνα, η φύλαξη των συνόρων, υπόθηκαν όλα αυτά και εσείς ήδη και όλα αυτά. Ε, κάθε φορά που ενσαρκώνουν το ευρωπαϊκό ιδεώδες μας βρίσκουν σύμφωνους. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε και στη διορθωτική πολιτική και στις ενισχύσεις ε, μήπως υπάρχει χώρος να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα. Νομίζω θα υπήρχε. Αλλά και εσείς εδώ στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είστε αρκετά θαραλέοι για να πάρετε τις αντίστοιχες αποφάσεις μαζί με το Συμβούλιο. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορεί ο καθένας να έχει ως αφετηρία και σημείο εκκίνησης ε, ένα σταθερό πρέσιο, με ε, ασφάλεια προγραμματισμού ε, για όλους τους κλάδους, για την υγεία, για την έρευνα, για τη γεωργία, για τη βιομηχανία, για το εμπόριο. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να βάλουμε τόσο ενθουσιασμό και τέτοια φόρα στη διεύρυνση των ιδίων πόρων και στην αύξηση των ιδίων πόρων. Είναι δύσκολο για ένα φορολογούμενο στην Ευρώπη, ο οποίος στενάζει από τις εισφορές και τους φόρους, να ε, απαιτηθεί μια επιπλέον προσπάθεια. Δηλαδή, μην αποθέτουμε τόσες πολλές ελπίδες στους ιδίους φόρους, Τουλάχιστον να τα αφήσουμε σε γενικές γραμμές όπως ήταν μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Οι εισηγητές μα κυρίω ο Ζεράρ είπε ότι αν είναι να υπάρξουν νέοι ήδη πόροι, νέοι φόροι α πούμε, τα εθνικά κοινοβούλια θα ψηφίσουν πρώτα. Και θα πρέπει, είπε, συγχρόνως να υπάρξει και μία ελάφρυνση άλλων φόρων, εθνικών ή τοπικών. Δηλαδή να μην υπάρξει επιβάρυνση φορολογική να υπάρξει εξορρόπηση. Ο κύριος Άγγελος Βόρτσης έχει τώρα το λόγο, παρακαλώ, από το Κυπριακό Κοινοβούλιο. Το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες δαπάνες για αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων, μετάβαση στη ψηφιακή ολοκλήρωση, προώθηση της αηφόρου ανάπτυξης, κλιματική αλλαγή, καινοτομία, μετανάστευση, αντιμετώπιση τη άνοδος του εθνικισμού και τη τρομοκρατίας. Πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικό, συμβάλλοντα στη βελτίωση της ποιότητα ζωή του Ευρωπαίου πολίτη, στη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνη των πολιτών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Θέλουμε να χαιρετήσουμε την προβλεπόμενη αύξηση των συνολικών δαπανών για το κεφάλαιο που αφορά την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, αύξηση κατά 15% σε πραγματικούς όρου, καθώς και των προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους. Τασόμαστε υπέρ της προτινόμενης ενίσχυσης της χρηματοδότησης για κάλυψη των νέων προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, διαχείριση εξωτερικών συνόρων, μετανάστευσης, ασύλου, ασφάλειας. Η κοινή αγροτική πολιτική και η πολιτική συνοχή θα πρέπει να παραμείνουν, κατά τη δική μα άποψη, ψηλά στι προτεραιότητε του νέου πολιετέ δημοσιονομικού πλαισίου 21-27, και να διατηρηθεί το επίπεδο χρηματοδότησή του στο νέο ε, πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων και προώθηση τη κοινωνική και οικονομική συνοχή ανάμεσα στα κράτη-μέλη τη Ένωση. Οι περιφερειακέ ανισότητε και οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών τη Ένωση, η Κύπρος είναι ένα νησί με γεωγραφικά απομονωμένη αγορά, πρέπει να ληφθούν υπόψη στου μελλοντικού σχεδιασμού τη ε, κοινή αγροτική πολιτική και τη πολιτική συνοχή. Η Κυπριακή Δημοκρατία, οφείλω να σα ενημερώσω ότι έχει επιφυλάξει ω προ την εισαγωγή των τριών προτινόμενων νέων ιδίων πόρων και ιδιαίτερα ω προ την εισαγωγή ίδιου πόρου που θα βασίζεται στην προτινόμενη κοινή ενοποιημένη βάση εταιρική φορολογία και το ύψο του προτινόμενου συντελεστή καταβολή, το οποίο ανέρχεται σε 3%. Αλήθεια, έχουμε προβληματιστεί ότι μπορεί η Μεγάλη Βρετανία να είναι εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση στι επόμενε χρονιέ που μιλάμε και θα είναι ενδεχομένω και ένα ισχυρό ανταγωνιστή. Πώ θα αντιμετωπιστεί αυτή η αύξηση του συντελεστή φορολογία κατά 3% σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα πλέον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος ως μικρό και απομονωμένο νησιωτικό, νησιωτικό κράτος, σε μια σταθή περιοχή με μεγάλες εξωτερικές προκλήσεις, διαθέτει περιορισμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία πρέπει να τύχουν σεβασμού από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιβολή εταιρικού φόρου πρέπει να παραμείνει αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, χωρί αυτό να εμποδίζει βεβαίω τη διασφάλιση τη άσκηση αυστηρότερου ελέγχου και βεβαίω μεγαλύτερη διαφάνεια για καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή. Σα ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το, λόγο στον συνάδελφο Κλάδιο Μπόργκη από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Monsieur you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκτίμησε ιδιαίτερα την ομιλία του κυρίου Ντεπρέ, διότι τόνισε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του αδιεξόδου αυτού. Τη σύγκρουση, δηλαδή, μεταξύ χωρών που είναι καθαρές, καθαροί και εκείνο που είναι καθαροί δικαιούχοι. Στην επιτροπή στην οποία ήμουν στο Ιταλικό Κοινοβούλιο, σε κάθε ακρόαση πάντα κάποιοι ζητούσαν αύξηση του προϋπολογισμού. στη γεωργία, αύξηση των πόρων για το α ή β τομέα. Και κάποιος σήκωνε το δάχτυλό του, το χέρι του τέλο πάντων, και έλεγε αν ζητήσουμε αύξηση, αν θέλουμε αύξηση του, του ευρωπαϊκού προπολογισμού και εφόσον εμείς είμαστε καθαροί πληρωτές, αυτό σημαίνει μείωση των δικών μας πόρων, διότι θα πληρώνουμε περισσότερα και θα παίρνουμε λιγότερα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, σκέφτηκε κάποιος ότι για τις χώρες της Ευρωζώνης, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημιουργήσε 3-3 με την διαδικασία ποσοτικής χαλάρωσης, 20 φορές τον προπολογισμό του του Ευρω... τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Τι θα είχε συμβεί από αυτά τα, αν από αυτά τα 3-3 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδινε ένα δις, ας πούμε, για, για νοσοκομεία, σχολεία, παράδεισος. Θα άνοιγαν οι ουρανοί, θα σάλπιζαν οι άγγελοι. Ξέρω ότι υπάρχει ο κανόνας ε, της μη χρηματοδότηση ενός κράτους μέλους, αλλά αν ήταν συλλογική η απόφαση, τι πρόβλημα θα υπήρχε αν είχαμε μια συμβολή από την ΕΚΤ στον κοινό προπολογισμό της Ένωσης. Κατά την άποψή μου θα μπορούσε να είναι μια λύση για να έχουμε περισσότερους πόρους και να μην χρειαστεί να επιβαρύνουμε τον προπολογισμό των κρατών μελών για να μετέχουμε σε αυτόν τον σημαντικό προπολογισμό της Ένωσης. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να έχουμε επιπλέον χρηματοδότηση και στην πράξη κανεί δεν πληρώνει, διότι το κόστο τη δημιουργία χρήματο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα προέρχεται από, από τον πληθωρισμό και τώρα δεν έχουμε πληθωρισμό. Άρα μπορούμε να, κάνουμε, να τα σκεφτούμε λίγο διαφορετικά από αυτά που τα σκεφτόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κυρία Μαρία Δελμάρ Άγγουλο, που είναι μέλος της Ισπανικής Γερουσίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συζητούμε για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και συμφωνούμε ότι θα πρέπει ο προπολογισμό να στραφεί στις βασικές μας προτεραιότητες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μας πρόκληση και θα είναι και η μεγαλύτερη μας συνεισφορά στην οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό είναι το θέμα της συζήτησή μας. Θα ήθελα εγώ να σας μιλήσω για μια σημαντική πρόκληση που νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε όλοι και που θα πρέπει να φαίνεται και ως προτεραιότητα στον προπολογισμό. Και αυτή είναι η δημογραφική πρόκληση, η υπογεννητικότητα, γύρανση του πληθυσμού, ε, μετανάστευση, αλλά και ανακατανομή ε, του πληθυσμού. Ε, σε πολλά μέρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ισπανία βλέπουμε ένα φαινόμενο απώλειας πληθυσμού, κυρίως στην Ήπεθρο. Άρα είναι σημαντική απάντηση που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η δημογραφική πρόκληση είναι πρόκληση για τις ίδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει σημαία της την ε, εδαφική συνοχή, την κοινωνική συνοχή και τελικά την ισότητα των ευκαιριών που θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Κατανοώ λοιπόν ότι έχει σημασία η Ευρώπη να δίνει απαντήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι στο περιθώριο, αλλά να ασχοληθεί και δημοσιονομικά με το φαινόμενο αυτό, γιατί σας είπα είναι από τι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Ε, πρώτο αυτό. Δεύτερο, έχει σημασία να πάρουν μέτρα τα κράτη-μέλη. Και παίρνουν μέτρα. Τώρα ε, ε, το συζητάει αυτό και η κυβέρνηση, αλλά και οι περιφερειακές και τοπικές η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να αξιολογήσει την απάντηση που δίνουν τα διάφορα κράτη-μέλη σε αυτή την πρόκληση για να δούμε πώς θα καταπολεμήσουμε την ερήμωση της υπαίθρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πάρει συγκεκριμένα μέτρα που να έχουν και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και πολύ σημαντικέ συνέργειε. Για να τελειώνω, το σημαντικότερο είναι ότι δεν είναι μόνο πρόκληση, ε, είναι και ευκαιρία αυτό το δημογραφικό. Ε, δεν πρόκειται για δαπάνες, για έξοδα, είναι και επενδύσεις αυτά, νέες δυνατότητες ε, απασχόλησης. Εκεί που είναι πιο γυραιός ο πληθυσμός χρειάζεται μεγαλύτερη φροντίδα, ας πούμε. Άρα έχουμε και ευκαιρίες για απασχόληση καινούριε και με την ψηφιοποίηση στην Ήπεθρο να φτάσει το διαδίκτυο στην Ήπεθρο, αυτό δημιουργεί και πλούτο και προστιθέμενη αξία σε πολλές περιοχές. Και νομίζω ότι βοηθώντας ε, τις περιφέρειες που δυσκολεύονται περισσότερο, τους δίνουμε ευκαιρίες. Γιατί η μεγαλύτερη ανάπτυξη δεν είναι μόνο ένα βήμα προς την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, όπως σας έλεγα, αλλά είναι και ένας σημαντικός παράγων για την οικονομική τους ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Παρτολομέ Προβλεύσκη και ελπίζω να πρόφερα σωστά το όνομά σας, είναι βουλευτής ε, στο Πολωνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Πολωνία στηρίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχουμε έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2021-2027 ε, σαφώς και χρειαζόμαστε τα κατάλληλα κονδύλια για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις προτεραιότητές μας αφενός, αλλά από την άλλη για να διατηρήσουμε και το σωστό επίπεδο χρηματοδότησης για τις πολιτικές που έχουν λειτουργήσει καλά τα τελευταία χρόνια. Η κοινή γεωργική πολιτική, για παράδειγμα. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, πιστεύω και πιστεύω ότι αυτό το πιστεύουν και πολλοί Πολωνοί, οι προτάσεις για περικοπές στην πολιτική συνοχή και την κοινή γεωργική πολιτική πάνε πολύ μακριά. Πιστεύω ότι θα έπληταν κυρίως στις λιγότερο πλούσιες χώρες και περιφέρειες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ως επιτοπλίστων. Πιστεύω ότι η οικονομική σύγκληση και η σύγκληση όσον αφορά τις υποδομές είναι κάτι που πρέπει να αναπτυχθεί στην Ευρώπη. Και η κατάλληλη θεραπεία μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η πολιτική συνοχής. Κάτι άλλο που πιστεύω και ξέρω ότι είναι κάτι που πιστεύει ο κόσμος στην Πολωνία και το στηρίζει, είναι ότι θα ήταν σημαντικό να υπάρχουν ε, οι άμεσες ενισχύσεις με περισσότερη ισορροπία επί ίσης όρης για όλους τους αγρότες ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το λέω γιατί πιστεύω ότι όλοι οι γεωργοί προσπαθούν να έχουν καλές προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος ε, και τα λοιπά, οπότε και οι άμεσες ενισχύσεις θα μπορούσαν να ήταν ε, αντίστοιχες. Εμείς πιστεύουμε ότι για ορισμένες χώρες που βρίσκονται λίγα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για πολλά χρόνια δεν είχαν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν όπως εκείνες της Δυτικής Ευρώπης, οι απαιτήσει για περιβαλλοντική προστασία της πλήττουν περισσότερο. Τώρα όσον αφορά τους ίδιους σπόρους, εμείς είμαστε υπέρ του φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και ίσως και υπέρ της φορολόγησης μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Και κάτι ακόμα. Για μας είναι μια πρόκληση, πρόταση για αλλαγές ε, στις χώρες εκείνες που βασίζονται στον άνθρακα. Οπότε είμαστε υπέρ της εξή πρότασης. Να υπάρξει ένα ξεχωριστό ταμείο αλληλεγγύης για την ενεργειακή μετάβαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Ο συνάδελφος τώρα από το Φιλανδικό Κοινοβούλιο, ο κ. Χάμακη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αλλαγή του κλίματος είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της εποχής μας. Ίσως θα μπορέσουμε να συνδέσουμε το πι δέλτα πι και την αλλαγή του κλίματος λύνοντας και τα δύο ζητήματα. Αν ε, έχουμε ένα είδος φόρο κλίματος θα μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα παίρνοντας χρήματα από τις χώρες που θα ήθελαν να πληρώνουν για να μπορούν να ρηπάνουν. Αυτός ο κλιματικός φόρος θα μπορούσε να είναι χαμηλός στο ξεκίνημα και να ανεβαίνει σταδιακά. Εάν αυξάνουμε από χρόνο σε χρόνο την, ε, έναν φόρο κλίματος, μπορούμε να κατευθύνουμε της, ε, την πορεία της Ένωσης και να βοηθήσουμε έργα που θα αναπτύσσονται με μικρότερη ρήπανση, θα είναι φθηνότερα σε όλες τις χώρες και τελικά όλες οι χώρες θα κατορθώσουν να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, ενώ η Ένωση θα έχει μεγαλύτερα έσοδα. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις δύο προκλήσεις μαζί. Κάτι άλλο που ήθελα να θέσω είναι το γεγονό πω όταν η Φιλανδία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνθήκη προσχώρησης είχαμε τους, τις ίδιες ε, προϋποθέσεις με την ε, χρηματοδότηση σε όλη τη Φιλανδία και διαφορετικές στην Ανατολική Φιλανδία. Γιατί θέλαμε εκεί να διαφυλάξουμε την φύση, και να υποστηρίξουμε την Βόρεια, τη Λαπωνία και την Ανατολική Φιλανδία. Πέρυσι η χρονιά, η, η απόδοση της γεωργίας ήταν κακή γιατί η χρονιά ήταν ε, στεγνή και η απόδοση χαμηλή. Η γεωργία δεν λειτουργεί λοιπόν σωστά και θα ήταν σκόπιμο η ενίσχυση αυτή στο βορρά και την Ανατολή να γίνει μόνιμη και όχι, και όχι να πάψει όπως είχε προγραμματιστεί με το παρόν MFP, ΠΔΠ. Ευχαριστώ. Τώρα, η Κλόντια Μιούλερ από την Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή. Ευχαριστώ πολύ. Τι μας δείχνει η συζήτηση με μεγάλη σαφήνεια και πάλι ότι στο PDP πολλοί συνάδελφοι έχουν τη δική τους εθνική σκοπιά. Πώς χρηματοδοτείται, ποια πολιτική και πώς φωτίζεται. Ο καθένας με βάση τις προσωπικές του εμπειρίες και το κράτος μέλος του. Θα πρέπει όμως να αναρωτηθούμε ποια είναι τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς το βλέπουμε εμείς και ποιες προκλήσεις θέλουμε να ξεπεράσουμε με το PDP και ποιες επενδύσεις για το μέλλον θέλουμε να μοιραστούμε από Και θα συνεχίσω από εκεί που ε, σταμάτησε ο συνάδελφος από τη Φιλανδία. Η κλιματική αλλαγή είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Και τι θα κάνουμε, πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Αυτό θα πρέπει να βρίσκει σαφή αντανάκλαση στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Μπέργκεκερ ε, που μίλησε προηγουμένω. Βεβαίω, κάθε πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο συμβιβασμό είναι. Ε, συγκεράζει διάφορα συμφέροντα. Τα ακούσαμε και εδώ. Ενίσχυση τη γεωργία, περικοπέ στη γεωργία. Ενίσχυση τη έρευνα και ανάπτυξη, ε, αύξηση των δαπανών, ελάφρυνση των φορολογικών υποχρεώσεων ή περικοπές ε, στις συνεισφορέ. Εγώ τι πιστεύω. θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε για τον πραγματικό στόχο, πρώτα απ' όλα. Και μετά θα δούμε αν χρειάζεται αύξηση των εισόδων, γιατί τότε δεν θα είναι αυτή η αποφασιστική ερώτηση. Είναι τι στόχους έχουμε, φτάνουν τα λεφτά για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Εάν η απάντηση είναι αρνητική, τότε θα πρέπει και μόνο τότε να αυξήσουμε τα κονδύλια. Ευχαριστώ κύριε μου. Ο Τζον Λάχαρτ από την Ιρλανδική Βουλή. Να απαντήσω σε πολλά ερωτήματα και σε σχόλια συναδέλφων από μια Ιρλανδική οπτική για να ενισχύσουμε την κατανόηση της συνέπειας ε, του Brexit στην Ιρλανδική οικονομία. Θέλω να ευχαριστήσω τους Ευρωπαίους εταίρους για την συνεχιζόμενη υποστήριξή τους ε, στην, στο υποεξέλιξη χάος που συνιστά το Brexit. Ακόμα δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος ε, του Brexit, δεν ξέρουμε τι μορφή θα έχει. Καμία χώρα λοιπόν δεν επηρεάζεται περισσότερο από αυτή την αβεβαιότητα από τη δική μου. Ιδίω γιατί δεν έχει κανένα έλεγχο της, των εξελίξεων στο σημείο αυτό. Όπως ξέρετε είμαστε χώρα με χερσαία σύνορα με το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτα γιατί δύο χρόνια μετά ακόμα δεν υπάρχει καμία εικόνα του ποιο μοντέλο Brexit θέλει να συμφωνήσει η κυρία Μέη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιπτώσεις και ο αντίκτυπος λοιπόν του Brexit είναι στην κορυφή της, της ατζέντα μας. Συμφωνώ και με του, τους προηγούμενους ομιλητές όπως αυτόν από την, το συνέδριο από την Φιλανδία και τη συνάδελφο από την ε, Γερμανία για το θέμα της αλλαγής του κλίματος. Από πέρυσι πολλές διεθνείς διασκέψεις υπογράμμισαν πόσο επίγον γίνεται το ζήτημα. Σε συνδυασμό με το θέμα της αλλαγής του κλίματος είναι και η διαγενειακή δικαιοσύνη τα παιδιά και τα εγγόνια μας, έχουμε, στα οποία έχουμε ευθύνη, για τα οποία έχουμε ευθύνη, θέλουν από μας να υπάρξουν δίκαια μέτρα για την αντιμετώπιση του κλίματος κάτω από το οποίο θα ζουν. Η Ιρλανδία έχει υιοθετήσει μια σειρά τέτοιων μέτρων που έχουν στόχο να μην πλήττονται οι πλέον ευάλωτοι, αλλά να τους χορηγούνται κίνητρα. Επίσης, με εντυπωσιάζει η ανάγκη της ενίσχυσης των, της εξουσίας των γυναικών σε πολλές χώρες, ακόμα και σήμερα οι γυναίκες δεν μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν όσο θα μπορούσαν να αποδώσουν. Τέλος, Εγώ πάντα συνεχίζω να πιστεύω σαν ε, πραγματικά ε, πεπισμένος ευρωπαϊστής ότι πρέπει να εμείνουμε στις αρχές της αλληλεγγύης και της αντιμετώπισης του εθνικισμού. Δεν πρέπει όμως να ενισχύουμε μέτρα Πρέπει να ενισχύουμε μέτρα που να δείχνουν τον ευγενή στόχο της συνένωσης των εθνών της Ευρώπης. Λίγα στην αρχή και όλο και περισσότερα. Αυτό νομίζω πρέπει να κατευθύνει τον στόχο μας. Τελευταίος ομιλητής, ο Τόκο Άλτο από το Φιλανδικό Κοινοβούλιο. Πρόεδρε, Ευχαριστώ για τις εξαιρετικές παρεμβάσεις όλων των συναδέλφων. Θέλω να σχολιάσω κάποια θέματα. Κόστος του Brexit. 30 δις υπολογίζεται. Τα εισοδήματα όλων, το, τα, έσοδα της Ένωσης θα μειωθούν, τα έξοδα θα αυξηθούν, άρα χρειάζεται νέες πηγές χρηματοδότησης όπως είπε και ο συνάδελφος από τη Φιλανδία, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ένα φόρο, ένα τέλος κλίματος. Εάν η Ευρώπη μπορέσει να, να φορολογήσει τις εκπομπές, θα μπορούσαμε ταυτόχρονα και να μειώσουμε τις εκπομπές και την εξάρτησή μας από ορυκτό, ενέργεια και ταυτόχρονα να αυξήσουμε τα κονδύλια της Ένωσης. Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με την ικανότητα προετοιμασίας όλων μας. Όπως ξέρουμε, η αλλαγή του κλίματος θα επηρεάσει τους πάντες. Πολλά μέρη του κόσμου και της Ευρώπης θα επηρεαστούν. Μπορεί να φτωχύνουν, η γεωργία, για παράδειγμα, θα πρέπει να αλλάξει λόγω της αλλαγής του κλίματος. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την φτώχεια των γεωργών Αλλιώ θα χρειαστεί εν τέλει να, να πληρώνουμε περισσότερα. Πιστεύετε ότι θα υπάρχουν κάποια πιο εύλογα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την, την αλλαγή του κλίματος. και που θα μας επιτρέπουν και να βρούμε και να χτυπήσουμε την ε, επιδείνωση του κλίματος και να βρούμε νέους πόρους για την Ένωση. Κοιτάξτε, είναι 7 παρατέταρτο, πρέπει να εγκαταλείψουμε στις 7 την αίθουσα. Θα ακούσουμε τον κύριο Σορίν Λαζάρ που θα κλείσει την ε, συζήτηση, αλλά ίσως ε, υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις από τους εισηγητές μας. Θέλετε να λάβετε λόγο κύριε Ντεπρέ, κύριε Φερνάντες, ε, εντάχει. Πορτογαλικά θα σας τα πω. Οι αλλαγέ του κλίματος είναι μία από τις ανησυχίες που βλέπουμε στο πι δέλτα γιατί μιλάμε για 20% των πόρων προς τον στόχο αυτό. Και το 2030 θέλουμε να το φτάσουμε στο 30%. Όλα αυτά προέρχονται από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις παρεμβάσεις τους. Νομίζω ότι με τα Εθνικά Κοινοβούλια θα έχουμε γρηγορότερα συμφωνία από ότι με τα κράτη-μέλη. Παράδοξο αυτό. Επανέρχομαι στο ερώτημα που τέθηκε για τον Ευρωπαϊκό Φόρο. Δεν υπάρχουν Ευρωπαϊκοί Φόροι. Είναι ψέμα να, που το επικαλούνται οι λαϊκιστές. Θέλω να τονίσω κάτι. Την ανάγκη αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάγκη εδαφικής συνοχής. Η εδαφική συνοχή δεν σημαίνει, δεν είναι το ίδιο πράγμα με τη σύγκληση. Υπάρχουν χώρες όπου σύγκληση και συνοχή διαφοροποιούνται και τα δύο ωστόσο χρειάζονται για να λειτουργήσει η Ένωση. Κύριε Γκόρδια Σάβελ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, όντως, εμείς πολύ πιο εύκολα και γρήγορα θα συμφωνούσαμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια παρά με το Συμβούλιο. Αλλά ανάλογα με τον ομιλητή και την ε, καταγωγή του άλλαζαν και οι προτεραιότητες. Και εγώ μίλησα ε, το είχα σημειώσει μάλλον να μιλήσω για την κλιματική αλλαγή και στην πρωτομιλία μου, αλλά για λόγους χρονικούς το ξέχασα μετά και δεν τον έφερα. Έχουμε στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη όταν κάναμε το πλαίσιο το παλιό, ήταν η στρατηγική 2020. Τώρα δεν έχουμε μια αποκλειστική στρατηγική σχετική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε πάρει τους στόχους ε, της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Ε, στέκομαι σε αυτό που είπε μια συνάδελφος από την Πορτογαλία για τη στήριξη στα προγράμματα εθνικών μεταρρυθμίσεων και το μηχανισμό σταθερότητας. Αυτό είναι αύριο στην ημερησία διάταξη και θα έχουμε περισσότερο χρόνο να το συζητήσουμε. Ένα πρώτο σχόλιο από πλευράς μου. Είναι δύο προτάσεις επιτάπητος αυτή τη στιγμή, αλλά πόρο απέχουν από τις ε, πραγματικές ανάγκες που έχει μια πολιτική και δημοσιονομική ένωση στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Στρέφομαι τώρα στους συνεισηγητές μας για τους ιδίους πόρους, ο Γιάννος Λεβαντόφσκι. Καλά, δεν είσαι και υποχρεωμένο. Ναι. όχι, γρήγορα. Ε, ε τα όσα ακούσαμε ε, από τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, δεν ήταν πολύ αντιφατικά με τις δικές μας προτάσεις, ε, εκτός από το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού 1% ε, του ΑΕΠ των κρατών μελών ε, και από αυτό το 90% περίπου επιστρέφει στα κράτη-μέλη γιατί είναι πολύ μικρές οι διοικητικές δαπάνες. Είναι επενδυτικός ο προϋπολογισμός λέτε και γι' αυτό χρειάζεται προβλεψιμότητα. Αυτό είναι και καλό μήνυμα για τους ε, Γερμανούς συναδέλφους, ο προϋπολογισμός μας θα πρέπει να είναι ίσως κελισμένος. Δεν μπορούμε να δανειστούμε, δεν μπορούμε να έχουμε το ταμείο μείον. Θα πρέπει πάντα να είναι ισοσκελισμένο ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Από το 2014 όμω και εντεύθεν ε, έχουμε επιδοθεί στο εγχείρημα να έχουμε περισσότερες υποχρεώσεις με λιγότερα χρήματα. Δηλαδή για πρώτη φορά ο προπολογισμό στο PDP 14 με 20 ήταν λιγότερο από ότι το 7 με 13. Αλλά είναι μονόδρομος. Ε, πάντα ε, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεις που πάνε στις Βρυξέλλες. Και αυτό δεν είναι απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι απόφαση των κρατών μελών. Ότι ε, περιμένουν περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκχωρούν περισσότερες αρμοδιότητες είναι δύσκολο να πετύχει περισσότερα με λιγότερα χρήματα. Υπάρχουν και όρια. Και σε ό,τι αφορά τη φωνή από την Πορτογαλία ε, για την επέκταση των ευθυνών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, είναι ήδη αρκετά επίμαχα τα όσα κάνει η ΕΚΤΑ σε διάφορα κράτη-μέλη. Για διάφορα κράτη-μέλη. Ε, θα μπορούσε να βοηθήσει στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ευχαριστώ, Ζεράρ Τιπχέ. Ναι, σύντομα, Πρόεδρε. Θέλω να πω στους συναδέρφους οι οποίοι ζήτησαν φόρο στα σύνορα για τα προϊόντα που δεν έχουν κάνει αρκετή προσπάθεια. Αν διαβάσετε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή της Κομισιόν, του Κοινοβουλίου, θα δείτε ότι αναφέρεται στην πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δύο λόγια επίση για τους καθαρούς εισφορεί. Πρέπει να κάνουμε μια μελέτη στην Ευρώπη. Γιατί δεν είναι απλώ αυτός που πληρώνει περισσότερα, είναι ποιοι εποφελούνται περισσότερο από το ευρωπαϊκό σύστημα και από την μεγάλη αγορά. Δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και λυπάμαι που το λέω, αλλά θέλω να το πω και να το ξαναπώ ξεκάθαρα, γιατί δεν πρέπει να λειτουργούμε σαν λογιστές απλώς και μόνο, αλλά να εκτιμήσουμε τα θετικά που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν καθίσουμε και αξιολογήσουμε ποιοι υποφελούνται περισσότερο από την ενή αγορά, θα δούμε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες από αυτές που είναι καθαρί φορές που υποφελούνται περισσότερο από την ενή αγορά. Είναι μια επιχρωματολογία που πρέπει να καταλάβουμε. Τέλος, τον Ιταλό συνάδελφο. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Γιάννου δηλαδή για την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι βασική αρχή αυτή η αυτονομία. Όταν ε, είχαμε την ποσοτική χαλάρωση, θυμόσαστε τι δύσκολες συζητήσεις έγιναν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οι πολιτικοί δεν παρεμβαίνουν. Μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε την τράπεζα με το σημερινό καθεστώς να ε, κάνει το ένα ή το άλλο. Όμως, στο έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δείτε ότι υπάρχει ένα παραθυράκι, γιατί μιλάμε για το περίφημο σενιοριάζ, δηλαδή για την δυνατότητα δυνατότητα όποιος υποφελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα κέρδη να μπορούν να χρηματοδοτήσουν ένα νέο μηχανισμό σταθερότητας. Δεν λέω ότι αυτό είναι ακριβώς αυτό που λέτε, αλλά είναι πάντως ένας προϋπολο... ένα... μια κατεύθυνση. Πολύ καλή ιδέα αυτή. Αλλά αυτά τα δικαιώματα σημαίνει μερίσματα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στους μετόχους. Οι μέτοχοι είναι οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Οπότε έχουμε να κάνουμε συγκοινωνούντα δοχεία εδώ, έτσι. Λοιπόν, βρήκα αυτή την ανταλλαγή απόψεων πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ πλούσια και ευχαριστώ πολύ όλους τους συμμετέχοντες. Αυτό που μας απασχολεί εμάς είναι να δείξουμε ότι αν οι χώρες πληρώνουν στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπάρχει προστιθέμενη αξία. Και μερικές φορές είναι δύσκολο αυτή την προστιθέμενη αξία να την υπολογίσουμε. Ευρώπη επίσης είναι αλληλεγγύη και μερικές φορές έχουμε την αίσθηση ότι παραμένει ε, πρόσθεση εθνικών εγωισμών και τίποτα άλλο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε από την Ευρώπη. Γιατί εδώ πέρα δεσμευόμαστε από το 2021 μέχρι το 2027 με αυτό το πολιτές πλαίσιο. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο ευελιξίας. Γιατί ας έχουμε υπόψη μας την Κίνα, τις Ηνωμένε Πολιτείες. Αλλιώς μπορεί με να τις έχουμε υπόψη μας, αλλά δεν θα έχουμε τα μέσα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις χώρες. Λοιπόν, Πρόεδρε, εσείς τώρα. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα και προσωπικά και εξ ονόματος της ε, ε, Ρωμανικής Προεδρίας και των Ρουμάνων συναδέλφων για τη διεξαγωγή αυτή της κοινοβουλευτικής εβδομάδας και για την παρούσα συνεδρίαση. Και φέτος είναι πολύ σημαντική αυτή η κοινοβουλευτική εβδομάδα για όλους μας. Ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, βουλευτές, ευρωβουλευτές για τη συνεισφορά και τις τοποθετήσεις τους για το τόσο σημαντικό αυτό θέμα, σημαντικό και για μας και για τους πολίτες. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Ταυτόχρονα είναι και βασικό μέλημα αυτό και ε, της ε, Ρουμανικής Προεδρίας μαζί με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα κατά τη διάρκεια ε, της Προεδρίας μας θέλουμε να ε, προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Φυσικά δεν υπάρχει, δεν νοείται πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο χωρίς ιδίους σπόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σήμερα ακούσαμε πολλά σχόλια, ένα ευρύ φάσμα επιχειρημάτων, τοποθετήσεων. Ε, το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτεί τις σημαντικότερες προτεραιότητες ε, για να έρονται ε, οι ε, ανισότητες μεταξύ των διαφορών κρατών και περιφερειών. Θα πρέπει να έχουμε οικονομική ανάπτυξη και νέες δυνατότητες να συνεχίσουν αυτές οι επιτυχημένες ιστορίες, success story που είναι η πολιτική συνοχής και η περιφερειακή πολιτική, αλλά και η κοινή γεωργική πολιτική, επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες, στην Ήπεθρο, ε, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις νέες αρμοδιότητες. Όλα αυτά είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικά. Ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για το διάστημα 2021-2027 θα πρέπει να εφαρμόζει την πολιτική συνοχής με τρόπο ευφυή. Δηλαδή τη δέσμευσή μας για μια Ευρώπη βιώσιμη ε, με ανάπτυξη. Έχω την τιμή να διαπιστώσω ότι πολλοί συνάδελφοι ε, τα βλέπουν αντίστοιχα τα πράγματα. Γι' αυτό πραγματικά ε, με βοηθάει να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου ως βουλευτής. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ βορρά, νότου, ανατολής, δύσης, αλλά όλα αυτά λύνονται και ε, διορθώνονται για να αντιμετωπίσουμε ε, καλύτερα το λαϊκισμό και να ε, το απαντήσουμε με τρόπο αποφασιστικό και στεναρό. Τι γίνεται με τους ιδίους πόρους, πώς θα δημιουργηθούν αυτοί, από πού θα προκύψουν. Δεν ξέρω ε, αν υπάρξουν νέοι φόροι ή νέες προσπάθειες φορολογικές. Ε, γίνεται λόγος για ένα νέο φόρο για τα πλαστικά που θα πρέπει να εισεχθεί. Όλα αυτά είναι σημαντικά βήματα ε, και φιλόδοξα που χρειάζονται τη χρηματοδότησή τους. Οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε υπερφορολόγηση των Ευρωπαίων πολιτών. Το αντίθετο. Θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη φορολογία έτσι ώστε όλοι οι πολίτες μας σε όλα τα κράτη-μέλη να αισθάνονται ότι είναι δική τους υπόθεση η Ευρώπη και όχι ότι οι ίδιοι βρίσκονται στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνθήκη των Παρισίων για το κλίμα. Ε, άρα μέχρι το 2027 θα πρέπει τουλάχιστον ε, το 25% να έχει γίνει ως προς τη μείωση ενώ των ε, εκπομπών καυσαέριων και διοξιδίου του άνθρακα. Ακούσαμε πολλές απόψεις, ακούσαμε πολλά επιχειρήματα και μάθαμε και πολλές εθνικές ιδιαιτερότητες. Πολλοί από τους συναδέλφους που μίλησαν, μίλησαν και προηγουμένως στην Ολομέλεια. Ελπίζουμε λοιπόν αυτά που ακούσαμε και προηγουμένως στην Ολομέλεια για την ε, πολιτική συνοχή, για την ανάπτυξη των περιφερειών, θα είναι πολιτικές που θα συνεχιστούν, γιατί πέτυχαν αυτές οι πολιτικές. Από τη Γερμανία ε, μίλησε κάποιος ε, για κριτήρια, για το πώς θα μετρήσουμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία πριν ε, προχωρήσουμε στα κεφάλαια ε, του προϋπολογισμού ε, του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Πολύ ωραία ιδέα. Φυσικά, πρώτα πρέπει να συζητήσεις για τους στόχους και μετά για τα οικονομικά. Κάθε ευρώ που επενδύεται θα πρέπει να πιάνει τόπο πέρα από την κάστοτε επένδυση, την επιμέρους. Πολύ σημαντικό. Ένα συνάδελφος από την Πολωνία είπε ότι οι εισφορές και ε, οι φόροι για το περιβάλλον δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών μελών. Ε, η κατάσταση είναι περίπλοκη και τα προβλήματα επίσης ε, δεν είναι απλά. Αλλά πιστεύω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι πρόθυμα και έτοιμα να ακολουθήσουν το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και να το κάνουν να στεφθεί και αυτό με επιτυχία. Λοιπόν, θέλω να σας καλέσω σε μια εκδήλωση που θα γίνει για τα 20 χρόνια του ευρώ από τις 7 και 4 Ε, ε, στον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ε, πάρτε και τις αποσκευές σας, θα σας δείξουν το δρόμο. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση, η οποία μας έδειξε ότι οι Ευρωπαίοι βουλευτές ανησυχούν για το μέλλον, για τα θέματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες και σας ευχαριστώ και εξ ονόματος της Ρουμανικής Βουλής για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, οι κλητήρες περιμένουν έξω, θα σα συνοδεύσουν. Θα σας βοηθήσουν να φτάσετε στον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.